Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επίτρο, κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, έφυγε η Επίτροπος. Εν αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα καταρχήν να σας διαβάσω μερικά στοιχεία από την Συμβουλευτική Επιτροπή του Διεθνούς Συμβουλίου για την Εξερεύνηση των Θαλασσών για το ΧΑΛΗ. Λέει ότι το απόθεμα του το χελιών ήταν σε κρίσιμη φάση το 2012 και το ποσοστό, ο δείκτης ανανέωσης βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά σημεία, κάτω από 1% για τη Βόρεια Θάλασσα και εκτός της Βορείου Θαλάσσης ε, λιγότερο από 6,5% σε σχέση με την περίοδο 1960-1979. Οι επιστήμονες της ISIS λένε ότι χρειάζεται να αναλάβουμε κατεπηγόντως μέτρα γιατί όλοι οι ανθρωπογενείς λόγοι θυσιμότητας, ε, η υδρορύπανση, ε, και άλλοι παράγοντες επηρεάζουν την αναπαραγωγή των χελιών. Θα πρέπει να απαγορευτεί η αλλιεύση χελιού. Αν είχαμε κάποια πιο χαρισματικά είδη, όπως τόνο ή ξηφία, σίγουρα θα είχαμε ε, και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ ή και πολύ πιο έντονη δημόσια κατακραυγή. Αλλά το ευρωπαϊκό χέλι που έχει καταπληκτικό βιολογικό ε, κύκλο ζωή, γιατί γεννιέται και πεθαίνει στη θάλασσα των Σαργασών και περνάει από διάφορε μεταμορφώσει. Η αλόχελο, κίτρινο, χέλι, αμόχελο, μέχρι να φτάσει σε φάση ορίμανση. Ε, δεν χρήζει, φαίνεται όμω απαραίτητη προσοχή. Ο κανονισμό που εξετάζουμε και θα ψηφίσουμε αύριο ανάγεται στο 2007, όταν τα κράτη-μέλη μετά από πολλά χρόνια συζητήσεων κατέληξαν τελικά να αναλάβουν κάποια μέτρα για να περιοριστεί η εξαφάνιση του ευρωπαϊκού χελιού. Έχουμε μία δεκαετία που συνεχίζουμε τη συζήτηση και ο κανονισμός ισχύει εδώ και μία πενταετία. Καθ' όλη τη διάρκεια αυτή το απόθεμα του ευρωπαϊκού χελιού έχει ε, συνεχίσει να μειώνεται. Το 2012 η ISIS έκρουσε και πάλι το κόδωνα του κινδύνου. Η ανασύσταση, ο εμπλουτισμός ε, των αποθεμάτων που ε, ε, προτάθηκε ω μέτρο διατήρησης κατά πάσα πιθανότητα δεν θα συμβάλλει στην ανασύσταση του αποθέματος ευρωπαϊκού χελιού τουλάχιστον με σημαντικό τρόπο. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα γιατί πολλά κράτη-μέλη έχουν στηρίξει τα σχέδια ανασύστασης στον εμπλουτισμό. Βέβαια δεν εφαρμόζονται κατευθυντήριε γραμμές για την επιβίωση του ιαλόχελου ή συνθήκες προκειμένου να μπορέσει να επιστρέψει στα θάλασσα των σαργασών για να αναπαραχθεί. Δύο σημαντικά πράγματα τονίζονται από τον κανονισμό. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει έκθεση για την σημασία του εμπλωτισμού ω ε, μέτρο συντήρηση του αποθέματο. Επίση, ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει μια νέα νομοθετική πρόταση πριν τι αρχέ του Μαρτίου του επόμενου έτου, που με μεγάλη πιθανότητα θα πρέπει ε, να μπορεί να σώσει το ευρωπαϊκό χέλι. Ελπίζω ότι και το Συμβούλιο θα αντιληφθεί την ανάγκη υποβολή και εφαρμογή αυτού του κανονισμού και δεν θα θάψει αυτά τα θέματα μαζί με άλλα διαχειριστικά θέματα εξαιτία διαφορετική ερμηνεία των αλληλευτικών ικανοτήτων. Γιατί στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει κατανομή αλληλευτικών ικανοτήτων. Οπότε συχνά στην ψηφοφορία ε, ε, δεν λαμβάνεται υπόψη ανάγκη ε, σύντομης ε, μεγάλης πρόθεσης αυτού του θέματος. Γιατί ε, θα πρέπει να προωθήσουμε βιώσιμη αλεία και να επιβάλλουμε και εμπορικές κυρώσεις σε τρίτες χώρες που επιτρέπουν μη βιώσιμη αλεία, ιδιαίτερα του χελιού. Το ευρωπαϊκό χέλι μάλιστα έχει περιγραφεί ως ε, ιδιαίτερα απειλούμενο είδο και εμπίπτει στο, στη σύμβαση του ISIS ε, για το εμπόριο επαπειλούμενων ειδών. Ευχαριστώ τους συναδέλφους που με υποστήριξαν και με βοήθησαν στην έκθεση. Ελπίζω ε, η διαδικασία να προχωρήσει και είμαι βέβαιη ότι οι επερχόμενες γενιές δεν ε, θα καταλάβουν τη λογική μιας απλής νομικής ε, προσαρμογής ενός κανονισμού που έχει στα χέρια του το πεπρωμένο ενός ολόκληρου είδους. És most a bizottság nevében Damanaki asszonyi σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα η Επίτροπο Ζαβανάκη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την κυρία Λέβιν και τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής Αλίας. Όπως γνωρίζετε, στόχος της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ο κανονισμός αυτός να γίνει συμβανθός με τη συνθήκη σχετικά με τις κατεξουσιοδότηση πράξης. Η έκθεση συμφωνεί με τις περισσότερες από τις προτάσεις μας. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων στην Επιτροπή Αλίας υπήρξαν αμφιβολίες για το αν ο κανονισμός αυτός είναι αρκετά αποτελεσματικός στην προστασία αυτών των χελιών. Θέλω να ευχαριστήσω πάντως και την κυρία Λέβιν για τον τρόπο με τον οποίο επανέλαβε την ανησυχία της εδώ. Από ό,τι κατάλαβα εσείς θα θέλατε να υπάρξει μια πληρέστερη αναθεώρηση των κανόνων ξεπερνώντας την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Να επαναλάβω σήμερα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σαν στόχο την ανάκαμψη ε, των ε, αποθεμάτων χελιού στην Ευρώπη. Εσείς επιθυμείτε να προετοιμαστούμε με διαφορετικό τρόπο και γι' αυτό είπαμε ότι θα προχωρήσουμε και ήδη αυτή τη στιγμή αναλύουμε τις τελευταίες εκτιμήσεις του ISIS ε, της εφαρμογής των ε, σχεδίων ηλεκτρονικής διαχείρισης από τα κράτη-μέλη. Περιμένουμε επίσης και τον Νοέμβριο του 2013 τα αποτελέσματα για τα αποθέματα χελιού του ISIS. Αυτές οι γνωμοδοτήσεις θα περιλαμβάνουν επίσης ε, και επανεξέταση του κανονισμού ε, και το κατά πόσον είναι συμβατός με την αρχή της πρόληψης. Επί τη βάση όλων αυτών των επιστημονικών στοιχείων, πριν από το τέλος του 2013 θα αναφερθούμε στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για την εφαρμογή αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων προστασίας των χελιών. Επί τη βάση των εκθέσεων αυτών θα δούμε αν θα χρειαστεί να υπάρξουν τροποποιήσεις στον κανονισμό για να βελτιώσουμε τους ρυθμούς ανάκαμψης των χελιών. Θα ήθελα να διαβεβαιώσω όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι φυσικά υπέρ της επιβίωσης του συγκεκριμένου είδους και αλλιεύματος. Ευχαριστώ Επίτροπε εξ ονόματος τώρα των πολιτικών ομάδων. Κουν, Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη κυρία Επίτροπε, κυρία Νταμανάκη, αξιότιμη συνάδελφε Λεβίν. Πράγματι σήμερα στη συζήτηση το θέμα που μας ενδιαφέρει είναι η προσαρμογή στη συνθήκη της Λισαβόνας, κυρίως όσον αφορά τη μεταφορά ε, των κατεξουσιοδότηση ε, πράξεων και των εφαρμοστικών πράξεων από την Κομισιόν προφανώς. Αυτό βέβαια που μας ενδιαφέρει είναι ότι ε, όσον αφορά το ευρωπαϊκό χέλι, η βιομάζα του και ο ε, δείκτης ανανέωσης του δεν βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα που πρέπει να το εξετάσουμε όπως αναφέρει και ο κανονισμός 1100 του 1207 ε, του 2007 με σχετικά με την διαχείριση του χελιού. Πράγματι το 2007 ήταν καθοριστική σημασία στο γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το Συμβούλιο ε, εκπώνησαν απαγόρευση εξαγωγής χελιού έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η βιομάζα του χελιού μπορεί να βοηθήσει έτσι ώστε να γνωρίζουμε πόσα χέλια ε, περνάνε στις ε, θάλασσες ε, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς πολλαπλασιάζονται τα χέλια στα φυσικά τους ενδιαιτήματα. Όλοι γνωρίζουν ότι υπάρχει μια μαύρη αγορά. Πρέπει λοιπόν αυτή την απαγόρευση εξαγωγών να τη συνεχίσουμε με συνέπεια έτσι ώστε να μπορέσουμε στο μέλλον να βελτιώσουμε τον δίκτυο ανανέωσης του χελιού. Υπάρχουν προγράμματα διαχείρισης που ήδη εφαρμόζονται σε πολλά κράτη-μέλη και αυτά πρέπει να συνεχίσουμε να τα παρακολουθούμε. Και το ιαλόχελο μπορεί να πολλαπλασιαστεί ε, σε υδατοκαλλιέργειες και έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα έτσι ώστε τα χελιά να τοποθετούνται μετά σε εσωτερικές ε, θάλασσες, σε λιμνοθάλασσες για να μπορεί εκεί να γίνεται αλίευση. Νομίζω ότι θα ήταν λάθος ε, το να διακόψουμε την διάρκεια ζωής ε, του χελιού που είναι 25 χρόνια και να πούμε θέλουμε αλλαγή. Δίκιο έχει η κυρία Λεβίν ότι χρειαζόμαστε την αξιολόγηση μέχρι τις 31 ε, για να δούμε πώς ακριβώς προχωράει το πρόγραμμα διαχείρισης και μετά θα δούμε τι θα κάνουμε στο μέλλον. Ε, σας ευχαριστούμε. Τώρα εκ μέρους των σοσιαλιστών ο κύριος Νίλσεν έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πράγματι η αλίευση των χελιών ήταν πάρα πολύ εντατική και φτάσαμε τα αποθέματα σε εξαιρετικά χαμηλό απαράδεκτο επίπεδο, καταστροφικό θα έλεγα. Ξέρουμε ότι τα χέλια ζουν δεκαετίες και το θέμα είναι ότι θα πρέπει να πάρουμε όλα τα απαιτούμενα μέτρα για να διασφαλίσουμε την επιβίωση του είδους και την ανάκαμψη των αποθεμάτων. Αυτό θα απαιτήσει ε, ένα μίξ θα έλεγα και ε, ταχυτά των μέτρων επί τη βάση των επιστημονικών φυσικά συστάσεων και επίσης κάποιων μέτρων τα οποία θα στοχεύουν στη μακροπρόθεσμη ε, προσπάθεια επιβίωσης. τα μέτρα τα οποία προτείνονται σε εθελοντική βάση μπορεί να είναι ε, θεωρητικά πάρα πολύ χρήσιμα αλλά θα πρέπει να ελέγχονται με σωστό τρόπο, με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, έτσι ώστε να πετύχουμε την ανασύσταση των αποθεμάτων. Εμείς ζητήσαμε από την Επιτροπή μας να κάνει νέες προτάσεις επί τη βάση των τελευταίων ε, και πλέον σύγχρονων επιστημονικών ε, συστάσεων. Ελπίζω αυτό να βοηθήσει ε, τα αποθέματα του ευρωπαϊκού χελιού. Σας ευχαριστώ. Εκ μέρους τώρα των φιλελευθέρων, το λόγο έχει ο κύριος Γκάλαχερ για δυόμιση λεπτά. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Καταρχήν να ευχαριστήσω θερμά την Ιζαμπέλα Λέβιν για το έργο της, ε, γιατί είναι πολύ σημαντική αυτή η έκθεση ευθυγράμμισης. Αναφίβολα, το, το απόθεμα ευρωπαϊκού χελιού βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Το 2007 περιλήφθηκε στο παράρτημα της ΣΑΙΤΕΣ, το ευρωπαϊκό χέλι, και το 2009 ε, καταγράφηκε στον κόκκινο κατάλογο του Άγιου για τα είδη που απειλούνται. Και μάλιστα κανονισμό του 2007 απαιτεί, απαιτεί από τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν μεμονωμένα σχέδια διαχείριση προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι της ανασύσταση ε, του αποθέματο σε βιώσιμα επίπεδα. Θα δούμε τι σημαίνει βιώσιμο επίπεδο βέβαια. Και πολλά μέτρα ε, προτάθηκαν όπως ε, η μείωση της αλίας ή η χρήση της, του εμπλουτισμού. Ε, δυστυχώς το Ιρλανδικό Σχέδιο Διαχείρισης ε, προβλέψε ολοσχερή, διαχει... Ε, ολοσχερή απαγόρευση της αλίας του χελιού κάτι που φέρνει σε πολύ δυσμενή θέση και είναι πολύ άδικο για τους Ιρλανδούς ψαράδες γιατί δεν έλαβαν κανένα αντιστάθμισμα από την απώλεια της, της δραστηριότητάς τους. Επίσης, το ευρωπαϊκό χέλι, το, το απόθεμα της Ιλανδίας εχει έχει συνεχίσει παρόλα αυτά 2009-2011 και σημαντικοί αριθμοί χελιού έχουν ε, καταστραφεί από τον υδροελεκτρικό σταθμό του Σάνων παρά τις προσπάθειες που έγιναν ε, να, να βοηθήσουν τα χελιά να περάσουν πάνω από τις ε, τουρμπίνες βιώσιμη διαχείριση του αποθέματος είναι ε, το κατάλληλο μέτρο για την Ιρλανδία. Από το 1980 ξεκίνησε ένα πρόγραμμα εμπλουτισμού ε, όταν ε, είχαμε τις πρώτες αποδείξεις για τη μείωση του αποθέματος. Τελικά η ομάδα μου αποφάσισε να καταθέσει μία ενιαία τροπολογία που οριακά ιτήθηκε στην Αρμόδια Επιτροπή προκειμένου να βοηθήσουμε τους αλληλείς να διαφοροποιήσουν την αλία τους, ιδιαίτερα στα κράτη-μέλη που αποφάσισαν να απαγορεύσουν πλήρως την αλίευση χελιού. Τώρα το θέμα της βιωσιμότητας. Είτε μιλούμε για πελαγικά, βεθοπελαγικά είδη, για το χέλι ή για το σκουμπρί, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι στις 10 Ιουλίου στην Επιτροπή Αλίας η ε, Επίτροπος ανέλαβε την ευθύνη και υποσχέθηκε ότι θα αναλάβει τα κατάλληλα μέτρα σε ό,τι αφορά το βορειοανατολικό Ατλαντικό και ε, για το θέμα της ε, κοινοποίησης. Και δεν αναφέρομαι στη Ρέγκα, αλλά στο Σκουμπρί. Έπρεπε να έχει ληφθεί αυτή η απόφαση ε, και αν ε, η καθυστέρηση οφείλεται στι θερινέ διακοπέ, έχει περάσει πια το καλοκαίρι και δεν έχουμε ακούσει τίποτα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γι' αυτό. Ο κύριος Γκρομπάρτζικ τώρα έχει το λόγο από τους μεταρρυθμιστές και συντηρητικούς. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα εισαγωγικά να ευχαριστήσω θερμά την Ιζαμπέλ για την πολύ καλή και ισορροπημένη της έκθεση, καθώς και για την ε, ε, προθυμία της και το συνεργάσιμο πνεύμα της ε, στις διαπραγματεύσεις. Είναι σημαντικό να δούμε ποια είναι τα απειλούμενα είδη. Είναι δύο βασικά τα επιχειρήματα της εισηγήτριας. Καταρχήν ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχουν αρκετές ή αρκετά ποιοτικές επιστημονικές πληροφορίες ό,τι αφορά το, τη μείωση του αποθέματος του χελίου και του λόγους. Επίσης ε, δεν είναι αξιόπιστα τα στοιχεία εκφόρτωσης των χελιών γιατί τα στοιχεία που δίνουν τα κράτη-μέλη δεν ε, συνάδουν με τα στοιχεία που έχει η Ευρωστάτ. Υπάρχουν ε, πολλά ελλειπή στοιχεία λοιπόν και ως προς τις ποσοστώσεις και τις εκφορτώσεις που δηλώνουν τα κράτη-μέλη και ε, τα στοιχεία της Ευρωστάτ. Και επίσης δεν έχουμε στοιχεία για τα πραγματικά αποθέματα του ευρωπαϊκού χελιού. Υπάρχουν λοιπόν ε, πολλέ, πολύ άγνωστοι στοιχεία εδώ πέρα. Και θα πρέπει να δούμε και την απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Βαλτική Θάλασσα που αυξάνει τις ε, ελεκτικές ποσοστώσεις για τα πελαχικά είδη και έτσι οδηγεί σε εξολόθρευση των ε, οικοτόπων και διατημάτων στη Βαλτική και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το Μερλούκιο, ε, τα αποθέματα βρίσκονται σε πολύ κρίσιμα ε, επίπεδα. Ζητώ λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει μια αναθεώρηση, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την σωστή εξακρίβωση των στοιχείων της αλίας και της πραγματικής αλίευσης. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Γκούσταψον εκ μέρου ε, της ΓΚΟΕ. Κύριε Πρόεδρε, ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ε, πάρα πολύ καλή δουλειά που έγινε. Υπάρχουν και πολλοί μύθοι τελικά ε, κανείς δεν ήξερε από πού προέρχεται το χέλι ε, γιατί ε, κανείς δεν το είχε δει να γεννιέται αλλά εν πάση περιπτώσει εκείνο που γνωρίζουμε είναι ότι το χέλι έχει έναν πολύ περίπλοκο κύκλο ζωής γεννιέται πολύ μακριά από εδώ και κατ' ουσίαν είναι αδύνατο να εκθρέψει κανείς χέλια ανεξάρτητα από το κατά πόσον ε, το εκτρέφουμε ή το αλλιεύουμε το ψάρι, αυτό που είναι απαραίτητο είναι να υπάρχει συνεργασία. Και αυτό που έχει σημασία είναι να απαγορευτεί η ελίευση ε, χελιού μέχρι να ανασυσταθεί το απόθεμα. Αν δεν ληφθούν δραστικά μέτρα δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Κατά τα άλλα θεωρώ ότι υπάρχει κίνδυνο στο τέλος να μην έχουμε καθόλου χέλια. Και όπως είπε και η κυρία Λουβίν, σε τελική ανάλυση Πώς θα το εξηγήσουμε αυτό στις επόμενες γενιές, ότι κατ' ουσίαν μόνοι μας εξολοθρέψαμε τα χέλια. Και τώρα, εκ μέρους ε, το EFD, ο κύριος Μπέλντερ. Κύριε Πρόεδρε, Κάποτε το θέμα αυτό ήταν καθαρά τεχνικής φύσεως. Τώρα όμως ε, υπάρχει και συζήτηση για το περιεχόμενο. Και εφόσον συζητάμε για το περιεχόμενο, είναι απαραίτητο να υπάρχουν και τα κατάλληλα επιχειρήματα. Δεν θα βοηθήσει ε, το χέλι, το να μην αλλιεύεται πια αυτό ε, έχει διαπιστωθεί στην ε, Επιτροπή Ελίας το πρόβλημα είναι μηχανότρατες και νομίζω ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να μετατρέψουν τα λεπτικά σκάφη. Όπως ε, λέμε και εμείς χαρακτηριστικά στην πατρίδα μας, πρέπει να βοηθήσουμε τα χέλια να επιβιώσουν, ε, να <clears throat> μπορέσουν να περάσουν από την άλλη πλευρά του φράγματος. Τώρα πλέον υπάρχει απόλυτη διαφάνεια, υπάρχει έλεγχος και αυτό βοηθάει τα χέλια. Εφέτος ε, θα έχουμε 25.000 ε, χέλια που θα μπορούν αυτά να επιβιώσουν στη θάλασσα των Σαργασών και αυτό πρέπει να στηριχτεί ως ε, πρωτοβουλία. Κύριος Χάρτονγκ. Voorzitter, nadat de EU de zeevisserij kapot dreigt te maken met haar waanzinnige omzwaai richting een aanlandplicht Κύριε Πρόεδρε, είναι προφανές ότι υπάρχει πρόβλημα σε σχέση με την αηφορία όταν μιλάμε για την εκμετάλλευση των αποθεμάτων χελιών. Τώρα έχουμε μια συγκεκριμένη πρόταση από το Κοινοβούλιο η οποία μπορεί να βοηθήσει. Νομίζω ότι ενδιάμεσα οι αλληλείς θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητες και ικανότητες που έχουν για να βοηθήσουν στην επιβίωση των ειδών. Φοβάμαι ότι τα μέτρα τα οποία έχει λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν καταστρέψει την αλληλεία και τώρα έρχεται η Επιτροπή για να βοηθήσει υποτίθεται rij maar door mijn straatje heen. Dank u wel. Androver urat illeti a szó. Gracias, presidente. Evidentemente en este debate Ευχαριστώ. Νομίζω ότι στη συζήτηση μπερδεύουμε διαφορετικά πράγματα. Θεωρητικά έχουμε μία πρόταση τροποποίηση του κανονισμού για την ευθυγράμμιση των διατάξεων του κανονισμού στις νέες διατάξεις της συνθήκης Λισαβόνας και ιδιαίτερα στις νέες αρμοδιότητες Ευρωπαϊκής ε, ε, Επιτροπής ε, και την ύπαρξη των κατεξιοδότηση και των εκτελεστικών πράξεων. Ουσιαστικά θα πρέπει να τροποποιήσουμε κάποιε διατάξει του κανονισμού με βάση τα άθρα 290 και 291 τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μία έκθεση ω πρόσχημα για να κάνουμε κάτι διαφορετικό από αυτό που οφείλουμε και να θέσουμε και ουσιαστικά θέματα που όπω λέει η ανάλυση δεν είναι το αντικείμενο που μα ενδιαφέρει, μια και η τροποποίηση αφορά τεχνικά σημεία που είναι η ευθυγράμμιση, κυρίω με τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Γιατί έτσι απομακρυνόμαστε από την κανονική η διαδικασία των τροπολογιών και διαφεύγουμε από την διαβούλευση που πρέπει να ισχύει πριν υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις προτάσεις στο Συμβούλο και το Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να τα έχουμε υπόψη όλα αυτά, γιατί όλοι καταβάλουμε τεράστιες προσπάθειες για να ευθυγραμμίσουμε τις νομοθεσίες μας στι συνθή, διατάξεις της Συνθήκης Λισαβόνας. Και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει η προσπάθεια αυτή να παρακτραπει προς άλλε. Τώρα, σε ό,τι αφορά το χέλι, είναι αλήθεια ότι το απόθεμα χελιού έχει μειωθεί κατά 95 έως 99% αν συγκρίνουμε τα τωρινά επίπεδα με τη δεκαετία του 80. Και αλήθεια είναι ότι η Διεθνή Ένωση για την Βράσπιση της Φύσης έχει χαρακτηρίσει το ευρωπαϊκό χέλι ως, είδο που, ως είδος που υφίσταται σημαντική απειλή. Επίση, το 2007 ο κανονισμό πρότεινε κάποια μέτρα για την ανασύσταση του αποθέματο και ζητά κυρίω από τα κράτη-μέλη να αναπτύξουν σχέδια διαχείριση προκειμένου να δημιουργηθεί τουλάχιστον 40% ε, της βιομάζας και να μπορέσει να ανασυσταθεί ε, το χέλι. Επίσης, η ΣΥΤΕ ε, λέει ότι το χέλι χρήζει ιδιαίτερη προστασία και θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα το θέμα της εισαγωγής και εξαγωγής. Αυτό αφορά το ευρωπαϊκό χέλι. Η κατάσταση του είναι κρίσιμη και θα πρέπει να δράσουμε. Αλλά ε, σήμερα το αντικείμενο δεν είναι το ευρωπαϊκό χέλι, αλλά η επιτροπολογία από ό,τι φαίνεται. Ευχαριστώ. Η κυρία Ρόντου έχει το λόγο. Πρόεδρε, ε, αγαπητή Μαρία Νταμανάκη, το ευρωπαϊκό χέλι τα πάει χάλια. Σας το λέω ξεκάθαρα. Ο κανονισμός για το χέλι έφτασε καθυστερημένα και τα κράτη-μέλη δεν τον εφάρμοσαν με ταχύτητα και ε, παράλληλα ε, μειωνόταν συνεχώς ε, το απόθεμα του χελιού. Σήμερα λοιπόν έχουμε το θέμα της προσαρμογής της συνθήκη της Λισαβόνας. Με την πρώτη ματιά αυτό μοιάζει να είναι μια βαρετή τυπολατρία αλλά δεν είναι έτσι γιατί πίσω από τη συνθήκη της Λισαβόνας ξέρετε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συναποφασίζει για την πολιτική αλίας. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τα αποθέματα θέματα του χελιού και ελπίζω τα προγράμματα να οδηγήσουν στην ανασύσταση των αποθεμάτων. Ε, Βεβαίω ε, δεν μπορούμε να προβούμε σε πιο ουσιαστικέ αξιολογήσει. Γι' αυτό λοιπόν εγώ στηρίζω τι συμβαστικέ ε, προτάσει που απαγορεύουν τα παρεπίπτοντα αλλιεύματα, όμως δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια μα στην πραγματικότητα και εάν κρυφτεί απαραίτητο να λάβουμε και άλλα μέτρα. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Στίβενσον. Ευχαριστώ πρόεδρε. Έχουμε δει μια κατάρρευση των αποθεμάτων χελιού κατά 90% και δεν είναι περίεργο γιατί τα σκοτώνουμε ε, σε όλες τις φάσεις της ζωής τους και εκεί που γεννιούνται ε, θεωρούνται μάλιστα και για ιατρικούς λόγους τα αλλιεύουν επίσης ε, και τα ενήλικα επίσης ψάρια και αυτά αλλιεύονται και τα φράγματα τα υδροηλεκτρικά δημιουργούν πάρα πολλά προβλήματα και δεν μπορούν να επιστρέψουν από το ταξίδι τους στη θάλασσα των Σαργασών. Νομίζω λοιπόν ότι ε, θα πρέπει να αναλάβουμε ταχύτατα δράση για να πάρουμε μέτρα που θα προστατεύσουν τα χέλια και γι' αυτό η έκθεση της κυρίας Λέβεν είναι εξαιρετική. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Καντέκ. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα Πολλοί παράγοντες επηρεάζουν ε, ε, τα αποθέματα των χελιών και η αλληλεία αλλά και οι, οι αποξηράνσεις ε, παραλιακών γεών όπως επίσης και τα υδροηλεκτρικά έργα. Όπως βλέπετε τα επιθετικά αυτά πράγματα είναι πάρα πολλά. Πρέπει λοιπόν να πάρουμε μέτρα. Παρ' όλα αυτά πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές και δεν θα πρέπει εμείς να προσπαθήσουμε να καταστήσουμε την αλληλεία από διοπομπαίο, από τράγο. Δεν νομίζω ότι η μείωση των αλλιευτικών δραστηριοτήτων είναι η μοναδική λύση. Ε, οι συγκεκριμένες περιοχές όπου ζουν τα χέλια πρέπει να ανασυσταθούν. Αλλά αυτό δεν προτείνεται από την έκθεση. Εμείς το ξεχνάμε. Στη Γαλλία, σαν παράδειγμα, η αλλιευτική κοινότητα έχει κάνει τεράστιες προσπάθειες για να μειώσει την θνητότητα αυτών των ειδών. Η παραγωγή ε, μικρών χελιών έχει μειωθεί σε σχέση ε, με το παρελθόν κατά 50-60%. Οι τα αλλιευτικά σκάφη έχουν επίσης μειωθεί πολύ. Πρέπει λοιπόν να μην αναθεωρήσουμε επιγόντως τον κανονισμό πριν έχουμε ε, την πλήρη κυκλοφορία των προγραμμάτων διαχείρισης του είδους. Θα πρέπει το Κοινοβούλιο να ε, περιοριστεί στην προσαρμογή στην Λισαβόνα, χωρίς περαιτέρω αλλαγές σε αυτή τη φάση. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα κυρία Τόμας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επιτροπέ, θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια και να πω ότι συμμερίζομαι τις ανησυχίες της για το απόθεμα του χελιού και την προστασία που χρήζει. Ε, δεδομένων βέβαια των στοιχείων που έχουμε βλέπουμε ότι κάποιες, ε, κάποια διεθνή επιστημονικά περίσματα δεν συνάδουν με κάποια ευρωπαϊκά ή με τη γνώμη των ε, αλλιέων. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε εξαντλητική αξιολόγηση των αποθεμάτων του χελιού σε όλα τα κράτη-μέλη. Και επειδή έχουμε καθυστερήσει στην παροχή στοιχείων από τα κράτη-μέλη, είναι απαραίτητο δυστυχώ να επιβάλλουμε κυρώσει στα κράτη-μέλη που είναι απρόθυμα σε συνεργασία ώστε να μην την πληρώσουν τελικά, να μην πληρώσουν τα σπασμένα ή το, το τίμημα της άγνοιας οι ίδιοι αλείς. Γιατί ήδη έχουν υποστεί τεράστιες θυσίες και πολλοί ασκούν με υποδειγματικό τρόπο την δραστηριότητά τους. Ας μην ξεχνάμε ότι σήμερα η θνησιμότητα χελιού κυρίως ρυθμίζεται από την αλή, ενώ ε, γνωρίζουμε ότι δεν οφείλεται η θνησιμότητα στην αλληλία αλλά περισσότερο στην ε, ρήπανση στην κατάσταση των υδάτων. Θα πρέπει λοιπόν να αναθεωρηθεί ο κανονισμό για την ανασύσταση του αποθέματο χελιού, λαμβάνοντα υπόψη ενημερωμένα στοιχεία πρόσφατα και να μην ε, συνδέει την θνησιμότητα μόνο με την Ελία. Θα πρέπει να εξασφαλίσει επίσημη αλυστική προσέγγιση και να λάβει υπόψη και τα συμφέροντα του κλάδου, εφαρμόζοντα σταθερά σχέδια διαχείριση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Νίκολσον τώρα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Στην ε, δική μου την περιφέρεια η ε, αλία χελιού είναι η μεγαλύτερη της Ευρώπης. Ε, έχουμε συνεταιρισμό των αλιαίων. Πάνω από 300 οικογένειες εξαρτώνται από αυτή την αλία και γι' αυτό πρέπει να προστατεύσουμε την αλία αυτή οι μέθοδοι ανασύστασης ε, του χελιού υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια και από το 1944 ο συνεταιρισμός έχει επενδύσει περίπου 5 εκατομμύρια λίρες για την ε, ανασύσταση του ε, αποθέματος. Τα χέλια λοιπόν του Λοχνέ πραγματικά αυτή τη στιγμή έχουν ένα πολύ καλό καθεζό. Πάντως δεν νομίζω ότι αυτή είναι, αυτό είναι μέρος της λύσης, ούτε ίσως και του προβλήματος. Επίσης θα πρέπει να υπάρξει μια εκτίμηση, μια αξιολόγηση πάνω σε ε, επιστημονικά δεδομένα. Εγώ ανέκαθεν υποστήριζα την κίνηση Επιτροπής προς την κατεύθυνση του να υπάρχουν υποχρεώσεις για την διαχείριση των χελιών. Ε, τα κράτη-μέλη πρέπει να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους ε, και να καταθέτουν ε, εκτέσεις που θα βοηθούν την Επιτροπή να προβαίνει σε αμερόληπτες αποφάσεις. Ευχαριστούμε πολύ και θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Φανίσε Ρόι. Κυρία Επίτροπε, κυρία Δαμανάκη, αυτό που θέλω να πω καταρχήν αφορά τις σχέσεις ε, των δύο οργάνων μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας. Και θέλω να πω το εξή ότι τώρα η συζήτηση είναι ουσιαστική. Το 90% του χελιού εξαφανίζεται και εμείς πρέπει να αναλάβουμε δράση. Οι άνθρωποι πλέον απευθύνονται σε εμά και μας στείλουν το θέμα και αν δούμε το τι εξάγεται γίνεται λόγος για λαθρεμπόριο ε, των ε, ιαλόχελων και άλλων ειδών χελιού. Κάτι λοιπόν δεν πάει καλά και αυτό οφείλεται στο ότι κανείς δεν τηρεί τις υποχρώσεις του. Γι' αυτό λοιπόν το Κοινοβούλιο δεν θέλει να έχει κατεξουσιοδότηση πράξης. Εμείς επιθυμούμε να εμπλακούμε στην όλη υπόθεση έτσι ώστε αν κριθεί απαραίτητο να μπορούμε να επέμβουμε. Έγινε λόγος και για την Ολλανδία. Στην Ολλανδία γίνονται αρκετά. Υπάρχουν ε, προγράμματα διαχείρισης ε, χελιού και αυτές είναι δραστηριότητες ε, που αναπτύσσονται με υπευθυνότητα. Βεβαίως και είναι κερδοφόρες όλες αυτές οι δραστηριότητες. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες, αλλά όλα αυτά πρέπει να φτάσουν κοντά στον πολίτη. Και εγώ νομίζω έφερες με ένα παραδείγματα για το πώς μπορούμε να επιτύχουμε τους στόχους μας. Σας ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στην διαδικασία Catch the Eye. Κυρία Μέντελσον, ευχαριστώ στη δική μου εκλογική περιφέρεια στο Λόχνη. Έχουμε το καθεστώς PDI και δεν υπάρχει κάποια άλλη μορφή αλίας που έχει τέτοια διαχείριση. Περίπου 300 ε, οικογένειες στο Λόχνη εξαρτώνται από την ε, αλία χελιού και έχουμε στο Λόχνη την πιο βιώσιμη αλία χελιού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και φυσικά αναγνωρίζουμε την ανάγκη ε, διατήρησης του αποθέματος και ε, την εξασφάλιση βιώσιμης ε, αλίας και βιώσιμων ελευτικών πρακτικών. Ε, τα τελευταία δέκα χρόνια 5 εκατομμύρια αφιέρωσαν στην αγορά και εμπλουτισμό των ιαλόχελων και συμβάλλουν στην ανασύσταση του ευρωπαϊκού αποθέματος. Και μάλιστα σε συνεργασία με Ινστιτούτα Βιοεπιστήμης προσπαθούν να εκτιμήσουν την κατάσταση του αποθέματος. Αλλά δεν θέλουμε κάποια πρόταση που θα επηρεάζει τη, τους αλληλείς και τη δραστηριότητά τους αν δεν έχει προηγουμένως ολοκληρωθεί μελέτη επιπτώσεων που θα στηρίζεται σε ανεξάρτητη επιστημονική συμβουλή. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Φερέρα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η διαχείριση του αποθέματος ευρωπαϊκού χελιού αντιμετωπίζει μια τεράστια δυσκολία. Έχουμε ελάχιστα επιστημονικά στοιχεία και δεδομένα που να στηρίζουν αυτή τη διαχείριση. Ένα πρόβλημα που επιδεινώνεται από την ε, σημαντική ε, έλλειψη που έχουν χώρες όπως η Πορτογαλία και εκεί ε, δημόσια Ινστιτούτα δυστυχώς έχουν παραλύσει λόγω και της οικονομικής κρίσης. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο προς τι οι κανονισμοί αν δεν συνοδεύονται από πόρους και κονδύλια που θα μας επιτρέπουν να εφαρμόσουμε τα παρέτα μέτρα γιατί η απειλή κατά του ευρωπαϊκού χελιού στηρίζεται σε πολλούς παράγοντες που όλοι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Δεν μπορούν να πληρώνουν τα σπασμένα μόνο οι αλείς και αυτοί να βαρύνονται για την ανασύσταση του ευρωπαϊκού χελιού. Γιατί η παράνομη αλία που δυστυχώς υπάρχει δημιουργεί τεράστια πίεση κρίση στο απόθεμα και γι' αυτό ε, και είναι καλύτερο να αντί να απαγορεύσουμε την αλία κίτρινόχελου θα πρέπει να επικεντρωθούμε στη διάσωση περισσότερο μεγαλύτερου ποσοστού του ιαλόχελου που είναι απαραίτητο για την αναπαραγωγή. Σας ευχαριστώ. Δεν ζητάει κανείς άλλο το λόγο στη διαδικασία του Catch the Eye. Οπότε μπορώ να ξαναδώσω το λόγο στην Επίτροπο, την κυρία Δαμανάκη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να επαναλάβω ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει σαν στόχο την σε εισαγωγικά λισαβονοποίηση της ρύθμισης. Αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε είναι να ευθυγραμμίσουμε την, τον υπάρχοντα κανονισμό στη νέα συνθήκη, στη συνθήκη της Λισαβόνας. Καταλαβαίνω βέβαια ότι είναι λογικό μια και έχουμε τόσες ενδείξεις ε, ότι τα αποθέματα δεν ε, βαίνουν καλώς, να εκφράζουν τις ανησυχίες τους τα μέλη του Κοινοβουλίου. Και σας είπα ότι τις ανησυχίες σας θα τις λάβουμε υπόψη. Αυτό το οποίο ήδη έχουμε κάνει είναι ότι έχουμε ζητήσει από τις επιστημονικές μας ε, υπηρεσίες να μας δώσουν τα απαιτούμενα στοιχεία. Ζητήσαμε επίσης και τα διαχειριστικά προγράμματα των κρατών μελών. Περιμένουμε λοιπόν να γίνει μια συνολική αξιολόγηση, θα αναλύσουμε τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης και όπως είπα πριν, μέχρι το τέλος του χρόνου θα επανέλθουμε ε, ε, και προς το Συμβούλιο με μια τελική αξιολόγηση για το τι κάνουμε και τι πρέπει να κάνουμε για να βελτιωθεί η κατάσταση των αποθεμάτων. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο τελικά στην εισηγήτρια. Ευχαριστώ και ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που έλαβαν μέρος στη συζήτηση και κυρίως που εξέφρασαν την υποστήριξή τους για την έκθεσή μου. Ευχαριστώ τους συναδέλφους που ανέφεραν και τους άλλους παράγοντες που απειλούν το απόθεμα ευρωπαϊκού χελιού, παρόλο που δεν το συζητήσαμε καθόλου αυτό το θέμα. Θα ήθελα όμως να υπογραμμίσω στα, στους ευρωβουλευτές από τη Βόρεια Ελλανδία το να χρησιμοποιούν το ε, νόρο βιώσιμο σε σχέση με το ευρωπαϊκό χελί είναι πολύ δύσκολο γιατί έχουμε μόνο ένα ενιαίο ευρωπαϊκό ε, απόθεμα χελιού Οπότε, παρόλο που μερικοί ελίες μπορούν να θεωρούν ότι ασκούν βιώσιμη αιλία, από τη στιγμή που έχουμε 99% μείωση του αποθέματος και δεν έχουμε κριτήρια ούτε παρακολούθηση των συνθήκων ανασύστασης ε, ή εμπλουτισμού, δεν μπορούμε να μιλούμε για βιώσιμη αιλία χελιού σήμερα. Αυτό που ζητούμε από την Επίτροπο είναι και μια αξιολόγηση του μέτρου του εμπλουτισμού, γιατί αυτό είναι κάτι το καινούριο. Θα πρέπει να αξιολογηθεί το κατά πόσο είναι χρήσιμο για τη συντήρηση. Γιατί δεν είμαστε σίγουροι ότι ο εμπλουτισμό συμβάλλει στην ανασύσταση του αποθέματο του Ευρωπαϊκού χελιού. Σε ό,τι αφορά την θρησιμότητα του χελιού κατά τη διάρκεια ε, τη αλίευση των μικρών ή ή κατά τη μεταφορά ή σε ό,τι αφορά τη μετάδοση των ασθενειών ή το κατά πόσο τα εμπλουτισμένα χέλια μπορούν να επιβιώσουν και μπορούν να κολυμπήσουν μέχρι τη θάλασσα των Σαργασών για να αναπαραχθούν και όχι απλώς ε, να αλλιευτούν στην πορεία. Μιλούμε για ευθυγράμμιση, αλλά πολλές φορές ε, είναι δύσκολο να είναι κανείς ε, συνεπής ακόμη και με, στην ομάδα του. Γιατί γνωρίζουμε ότι για, την, για το σχέδιο διαχείρισης Βαλτικής, το ΕΛΚ, τάχθηκε υπέρ κάποιων σημαντικών αλλαγών σε ό,τι αφορά την έκθεση λισαβονοποίησης. Δεν είναι λοιπόν ότι το Άλκιν είναι πάντα συνεπέ ε, στην υιοθέτηση των απόψεών του. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, κυρία Επιτρόπο γιατί φαίνεται ότι λαμβάνεται ότι η σοβαρότητα και το κατεπήγον της κατάστασης ε, απαιτεί κάποια επιπλέον στοιχεία στο σχέδιο ανασύσταση του Ευρωπαϊκού Αποθέματο Χελιού. Και σε όσους αναφέρθηκαν στην, στις παράνομες εξαγωγές του Ιαλόχελου. Ναι, ε, πολύ ευχαρίστω το κάνουμε, αλλά δεν είμαστε συνεπείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί από τη μια αναγνωρίζουμε ότι το ευρωπαϊκό χέλι βρίσκεται υπό εξαφάνιση και από απειλή γιατί θα πρέπει καν να εξαγάγεται και ταυτόχρονα είμαστε δυσακτικοί να ρυθμίσουμε το εμπόριο εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε συνεπείς, ιδιαίτερα μια εποχή που η Ευρωπαϊκή Ένωση σκέφτεται να επιβάλλει εμπορικέ κυρώσει σε βάρο ε, άλλων χωρών που ασκούν μη βιώσιμη αλεία. Θα πρέπει και εμεί να εφαρμόζουμε τι ίδιε προδιαγραφέ και να είμαστε το ίδιο απαιτητικοί και με του εαυτού μα. Σα ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε και εμείς. Ε, έτσι λοιπόν, ολοκληρώθηκε αυτή η συζήτηση. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο το μεσημέρι. Και το επόμενο θέμα στην ημερησία διάταξη είναι η έκθεση της